ο κύριος Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθίστε, λέει ο Προεδρεύων, κύριος Παπαδημούλης. Please call it, thank you. Σας παρακαλώ καθίστε. Πριν προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες, uh, Mr. Pitella asked